Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση όσον αφορά τις ερωτήσεις. Τα πρακτικά της, της ε, συνεδριάσεως θα υποβληθεί στην έγκριση του Κοινοβουλίου στην επόμενη σύνοδο. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα διαβιβάσω μέσω...